είναι, ε, θελοτυφλούμε και να δούμε ότι πολλά προβλήματα των ομάδων αυτών εξαρτώνται βασικά από αυτούς τους ίδιους. Τα προβλήματα των Ρωμά. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Οπότε πάμε στο επόμενο θέμα της μεσηδιάταξης. Έκθεση Φερνάντες για την κατάσταση των προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012. Τμήμα 1, Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή, στον κύριο Φερνάντες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν ε, στην σύνταξη της έκθεσης αυτής ε, και στη συζήτηση που προηγήθηκε. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους κοιόδης συζητητές όλων των πολιτικών ομάδων. Η έκθεση αυτή σημαίνει ότι το 2012, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έχουμε ένα προπολογισμό λιτότητας, ε, έλεγχος των δαπανών, αυστηρότητα, λιτότητα ουσιαστικά, γιατί σε σχέση με την αρχική πρόταση μειώθηκε το ποσό κατά 49-50 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε ευρία πλειοψηφία υπέρ της πρότασης αυτής ε, του Κοινοβουλίου. Και μάλιστα ξεπεράσαμε και αυτά που είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε. Είχαμε πει ότι να υπάρχει τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Ε, ε, αυτό βέβαια δεν τηρήθηκε, που σημαίνει ότι ο του 2012 συνεπάγεται περικοπές, μείωση των δαπανών. Και κάτω από το 20% του τίτλου 5, που αφορά δηλαδή τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάποια χρόνια δεν είχαμε φτάσει αυτήν την οροφή. Η διάσκεψη των Προέδρων Μας είχε θέσει ως στόχο το 20%, το 22% συγγνώμη. Δεν το φτάσαμε για φέτος αυτό το 22%. Το 2012 όμως πρέπει να κάνουμε και κάποιες οικονομίες. Με βάση την αρχή της χρηστής ε, διαχείρισης. και του σωστού υπολογισμού των δαπανών. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση για όλες τις δαπάνες θα υπάρχει ανάλυση κόστους ωφέλους για όλες τις δαπάνες. Και έτσι θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε περαιτέρω χρήματα και στη φάση της υλοποίησης. Νομίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια να κάνουν οικονομία. Το περιθώριο για τον τίτλο 5 διοικητικές δαπάνες για τα θεσμικά όργανα όπως είπα θα έχουμε κάποιο πλεόνασμα 190 εκατομμύρια ευρώ 100 εκατομμύρια ευρώ υποτίθεται ότι θα πρέπει να, που θα πήγαιναν στις διοικητικές δαπάνες θα πρέπει να μεταφερθούν για την νεολαία, στον τίτλο για την νεολαία. Γιατί εκεί. Γιατί σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες και υπάρχουν διπλάσια ποσοστά ανεργία μεταξύ των νέων σε σχέση με άλλε ηλικιακέ ομάδε. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Επίσης έχουμε τη στρατηγική του 2020 η νεολαία είναι προτεραιότητα και σε αυτή τη στρατηγική. Αν δούμε την εγκατάλειψη του σχολείου, αν δούμε την ε, πορεία των ε, αποφύτων του σχολείου, πόσοι έχουν ε, διπλώματα πανεπιστημίου, Βλέπουμε ότι αποτελούν προτεραιότητες, ε, η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα και δεν θα πρέπει τροπολογίες οι οποίες οδηγούν ε, σε λάθος ε, πορεία, δεν θα πρέπει να γίνουν δεκτές. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τώρα από το ΕΛΚ με του αγορητέ των διαφόρων ομάδων. Δίνουμε στον κύριο Ολμαέρ το λόγο για δύο λεπτά. Στην κυρία Ολμαέρ. Ο προπολογισμό για το 2012, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδρε, αντιμετωπίζει δυσκολίες γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Γι' αυτό χαίρομαι που καταφέραμε επί της αρχής να συμφωνήσουμε για τον προπολογισμό μας στο Κοινοβούλιο και ακολουθήσαμε την αρχή του να μην υπάρξουν έντονες ε, αυξήσεις και να λάβουμε υπόψη και τον ε, ποσοστό πληθωρισμού. Ο στόχος που ανέφερε ο συνάδελφος Φερνάντες για την νεολαία είναι πάρα πολύ σημαντικός και μας αφορά ιδιαίτερα εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να διατίθενται πιο πολλά χρήματα στην νεολαία από ό,τι συμβαίνει ως τώρα, γιατί στην τελική ανάλυση οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν ε, θέση απασχόληση, που θέλουν ιδιαίτερη ε, υποστήριξη θα πρέπει να λάβουν την υποστήριξη αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα επιπλέον 100 εκατομμύρια είναι πολύ θετική εξέλιξη. Και σε ό,τι αφορά τα κτίρια, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό σε θέματα στέγασης να υπάρξει μεγάλη αποδοτικότητα. Συγγνώμη, να υπάρξει μια μεγάλη αποβατικότητα προκειμένου να μετρηθεί η κατάσταση και να βελτιωθούν τα πράγματα από χρηματοδοτική άποψη. Θεωρώ ότι τα μέσα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει κατά τη διάρκεια του έτου να χρησιμοποιηθούν για να αποφύγουμε ενδεχόμενα επιτόκια προκειμένου να μην ξοδευτούν τελευταία στιγμή στον περίοδο του Δεκεμβρίου, όπως αποκαλείται τα χρήματα αυτά και προκειμένου να χρηματοδοτηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα κτίρια. Θα φροντίσουμε να ελέγχεται η αρχή της λειτουργίας και προκειμένου και στον τομέα της ε, οικοδόμησης να πληρούνται οι σωστές αρχές οι δημοσιονομικές. και να ακολουθούνται οι σχετικοί κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Βόγκαν για δυόμιση λεπτά. Κύριος Βόγκαν. Ευχαριστώ. Καταρχάς να αποτίσω φόρο τιμής προς την εισηγητή με τον τρόπο που προσέγγισε το προπολογισμό και την αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να αποφύγει μεγάλες αυξήσεις στις δαπάνες του για το 2012. Αυτό ισχύει όλο ιδιαίτερο, διότι ξέρουμε το Συμβούλιο προτίθεται να περικόψει τον προπολογισμό του κατά 4%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τον προπολογισμό τη κατά μόνο 1%. Η Επιτροπή των Περιφερειών κατά 2,9% και ο ΚΕ ε, κατά μικρότερο ποσό. Αρχική πρόταση που έγινε από το Προεδρείο, νομίζω, του 5,2% ήταν πολύ υψηλό. Η μείωση της αύξησης το 2,3% λοιπόν αποτελεί προόδο είναι μια περικοπή σε πραγματικούς όρους περίπου του 0,5%. Προσωπικά θα ήθελα να δω την αύξηση ακόμα μικρότερη και στο μέλλον πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο ούτω ώστε να εντοπίζουμε εξοικονομήσει στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Όμω θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι οικονομίε έχουν γίνει. Καλωσορίζω τι οικονομίε που έγιναν στην, προστεξολο... στη μονάδα αξιολόγηση προστιθέμενη αξία. Περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ εξοικονομήσαμε από εκεί. οικονομίε όσον αφορά τις εξατήσεις ενημέρωση, πολιτική ε, χαρτικά ε, και την πρόταση να μειωθεί το αποθεματικό για πήγους ανάγκε στα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Ε, όλα αυτά είναι πραγματικές οικονομίε του περίπου 13,7 εκατομμύρια ευρώ συν ε, την, ε, τις δαπάνες περικοπές που κάναμε η Λισαβόνα και η διεύρυνση και άλλε περικοπές θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά τελικά όμως κάναμε κάποιες οικονομίες. Έχω δύο σημαντικά θέματα που εκκρεμούν να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα η πρόταση των 100 εκατομμυρίων ευρώ από τα αποθέματα του κεφαλαίου 5 να πάνε στην πολιτική για την νεολαία, κάτι που περιέγραψε και ο συγητής. Στην τροπολογία μας μαζί με άλλες ομάδες, στην τροπολογία 7 είπαμε ότι αυτή η μεταφορά θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο όμως σύμφωνα με τις προτεραιότητες της γενικής, του Γενικού Προλογισμού του 2012. Άρα χρειάζεται συζήτηση το θέμα πριν να ληφθεί μια απόφαση εάν θα γίνει αυτό και πού θα πάνε τα χρήματα. Με άλλα λόγια, πού θα δαπανηθούν τα χρήματα εάν τελικά λάβει η χώρα μεταφορά. Είναι πολύ πρόημο τώρα να δεσμευθούμε. Δεύτερον, υπάρχει και το θέμα του οίκου ευρωπαϊκή ιστορία. Καλή ιδέα, πολύ καλή ιδέα, αν έχουμε πολλά χρήματα, αλλά τώρα δεν είναι σωστή στιγμή. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ε, επιχειρησιακό. Θα πρέπει να ακολουθηθεί ιδέουσα κοινοβουλευτική διαδικασία, ίσω μέσω κανονική διαδικασία του προπολογισμού αργότερα φέτο, ώστε να εκφράσουν την άποψή του οι βουλευτέ για το πρόγραμμα. Πάνω σε αυτό, Πρόεδρε, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και για άλλα θέματα, να ειδωθεί ότι λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις για τον προπολογισμό μας. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για το κοινό. Να φανεί αυτό. Σας ευχαριστώ για την Άλντε Αλβάρο για δύο λεπτά. κύριος Αλβάρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το έργο του εισηγητή ήταν καρποφόρο και αυτό καταδεικνύει ότι δεν είναι όλα τα χρήματα, δεν είναι τα πάντα τα χρήματα, αλλά χρειάζονται πάντα και χρήματα. Και η συζήτηση που γίνεται για το επίπεδο πληθωρισμού 2,5%, 2,7%, 2,3% δεν είναι τίποτα άλλο παρά ε, τσακωμός. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πού μπορούμε να κάνουμε οικονομία. συγκεκριμένα. Βασική προϋπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση και είναι σημαντικό η Γενική Γραμματεία αυτό να το πάρει σε σοβαρά η Επιτροπή Προπολογισμών να λαμβάνει όλα τα σχετικά τεκμήρια προκειμένου βάσει του σχεδίου προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσει πού μπορούν να γίνουν οικονομίες και πού υπάρχουν δυνατότητες οικονομία και όχι μόνο να λαμβάνει τις προτάσεις, τις τροποποιητικές της Γενικής Γραμματείας. Είναι μεγαλύτερος ο ρόλος μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπε και ο άδελφος ε, Φερνάντες, είχαμε αρκετές ευκαιρίες για 49 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που είπε, που δεν είπε, ότι θα πρέπει του χρόνου να αποφασίσουμε τι θα γίνει με τα κονδύλια αυτά που μεταφέρονται. Χαίρομαι για τις ε, οικονομίες. Χαίρομαι που καταφέραν να συνενωθούν οι μικρές ομάδες και να μας πείσουν εμάς τους μεγάλους ότι είναι σημαντικό να γίνουν τέτοιες οικονομίες σε διάφορους τομείς, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ιδρύματα κτλ. Ότι τέλος πάντων χαίρομαι που υπάρχει μια προσέγγιση για το πού μπορούν να γίνουν οικονομίες. Η συζήτηση για τα, για τα 100 εκατομμύρια ευρώ για την νεολαία είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορεί κανείς να αντιταχθεί. Ωστόσο να προσέξουμε, γιατί αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει με την έκθεση αυτή, θα πρέπει να ε, διαπραγματευτεί σε άλλες εκθέσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μας αποσπά την προσοχή από άλλα σημαντικά θέματα. Ωστόσο έγινε μια αρχή η οποία καταδεικνύει ότι δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα πιο πολλά χρήματα, αλλά χρειαζόμαστε τη δημοσιονομική πειθαρχία. Και νομίζω ότι κάνουμε ε, μια καλή αρχή σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους πρασίνους. Τρούπελ για μισή λεπτά. Κυρία Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σωστό στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλλει, να είναι πρόθυμο να συμβάλλει και να αυτοπεριοριστεί, να αυτοπιθαρχηθεί παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε φάση οικοδόμησης ε, του θεσμικού μας οργάνου και ότι λάβαμε νέες αρμοδιότητες με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι ήταν καλό και ορθό οι προτάσεις ε, του Προεδρείου που προέβλεπαν 5,2% περιορίστηκαν στο 2,5%. Αλλά να τονίσω ότι πρόκειται για ποσοστά κάτω από το όριο του πληθωρισμού. Μιλάμε για μείωση της αύξησης, όχι για πραγματική οικονομία. Να μην φοβόμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, Για τον ε, οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας να πω ότι επί της, η ομάδα, επί της η ομάδα μου θεωρεί ε, αυτή η υπηρεσία, ότι πρόκειται για μια υπηρεσία προς τους πολίτες. Αλλά χρειαζόμαστε και ένα business plan, προκειμένου όλοι οι όροι που διατυπώνονται να μπορούν να πληρούνται. Μόνο τότε μπορούμε να καταρτήσουμε ένα προϋπολογισμό με, αληθο... με ειλικρίνεια και αληθοφάνεια. Αν θέλουμε λοιπόν αυτή τη νέα προτεραιότητα που συνεπάγεται 60 εκατομμύρια επένδυση τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι, να πρόθυμοι να κάνουμε οικονομίες σε άλλους τομείς και όχι απλά να περιορίζουμε την αύξηση του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, θεωρούμε ότι στις πτήσεις ε, κάτω των τεσσάρων ώρων θα πρέπει να μην υπάρχουν ταξίδια στην ε, οικονομική κατηγορία business. Μία τελευταία πολιτική παρατήρηση για το πολιτικό τρίκ σε ό,τι αφορά τα 100 εκατομμύρια για την νεολαία. Φυσικά και εμείς οι πράσινοι θέλουμε να δώσουμε πιο πολλά χρήματα στη νεολαία. Α, α, αλλά αν αφαιρέσουμε αυτό το ποσό από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν χρηματοδοτούμε για παράδειγμα τα πολιτικά ιδρύματα και την υποπτία αυτών. Αυτό θέλουμε πραγματικά. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια εσφαλμένη απόφαση. Τα ιδρύματα αυτά χρειάζονται μια σωστή ρύθμιση. Θα πρέπει να έχουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες να λειτουργούν σωστά και θα πρέπει να διατεθούν τα κονδύλια για τους νέους ε, που τους αναλογούν. Νομίζω ότι αυτή ήταν η σωστή πολιτική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ για τους ειδικούς και μεταρρυθμιστές. Μπόκρος για 2,5 λεπτά. Κύριος Μπόκρος. Οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ενώσης ζουν μέσα σε μια σφαίρα αυταπάτης και παρεστήσεων. Το παράδειγμα το είδαμε σήμερα το πρωί. Οι ηγέτες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσης έλεγαν ότι η χρηματοστική κρίση είναι πίσω μας κατά πολύ. Τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια όπως αναφερόθηκε χθε σε άρθρο των Financial Times, έχει επιλογή Ευρώπη μεταξύ χρεοκοπία και βοήθεια για να τη γλιτώσει. Άρα χρειάζεται τεράστια, να απορροφηθεί τεράστια απώλεια. διαφορά μεταξύ των δύο είναι πώ τελικά διανέμεται η απώλεια. Στην περίπτωση τη χρεοκοπία, η γερμανικέ, οι γαλλική, οι ιταλικές, οι βρετανικέ τράπεζε και οι Γαλλικέ τράπεζε υποφέρουν και θα πληρώσουν οι μέτοχοι ε, τα λάθη, τα χρέη των Ιταλών, Πορτογάλων και Ελλήνων φορολογωμένων. Στην περίπτωση ε, οι Πορτογάλοι πολίτε, οι Έλληνε πολίτε και οι Ιρλανδοί πολίτε θα πληρώσουν στην περίπτωση προσπάθεια να γλιτώσουν οι τράπεζε. Άρα η προσπάθεια να αυξηθεί κατά 2,3% προπολογισμό ε, του Κοινοβουλίου είναι κάτι απαράδεκτο. Και θα πρέπει να πάμε πίσω στο 1% που είχε προτείνει ο Γιάννου Λεβαντόφσκι, ο Επίτροπο, για να δείξουμε μια αύξηση κάτω από τον πληθωρισμό ε, θα έδινε μεγάλη νομιμότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα μάτια των Ευρωπαίων ε, ψηφοφόρων. Δεν είναι μόνο το θέμα τη ανάπτυξη ε, και οι δομέ που μπορούν να αλλάξουν. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Όπω η Helga Triple ήδη είπε, δεν χρειαζόμαστε να ταξιδεύουμε business στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια πρόταση που προτείνουν οι πράσινοι, η ενωτική αριστερά και η ECR να μειωθούν τα οδηπορικά σημαντικά χρησιμοποιώντα ευέλικτα εισιτήρια οικόνομη σε περιπτώσει που η πτήση δεν είναι πάνω από 4 ώρε. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε για αριστερο στόλο μαύρων Mercedes Benz εδώ στο Στρασβούργο. Χρησιμοποιήστε το τραμ. Δεν χρειαζόμαστε το σπίτι τη ευρωπαϊκή ιστορία. Χάνει ανταγωνιστικότητα η Ευρώπη και γεωπολιτικό βάρο Άρα γίνεται ένα μουσείο έτσι κι αλλιώ. Υπάρχει τεράστια δυνατότητα οικονομιών όσον αφορά την ενέργεια. Τα γραφεία μα δεν έχουν θερμοστάτη και προσαρμοζόμενο ατομικό, σε ατομικό επίπεδο και εξοδεύουμε τεράστια ποσά ενέργεια κάθε χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε τεράστια οικονομίε στην ασφάλεια και στην πληροφορική. Και στι δύο περιπτώσει χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη υπηρεσία και πολύ λιγότερα χρήματα. Θα πρέπει να επεξετάσουμε και να θεωρήσουμε όλο και το κόστο τη υγειονομική περίθαλψη διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γενναιόδορη επιλογή υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητε αρνητικέ και θετικέ. Περί αυτού πρόκειται ο προπολογισμό. Υπάρχουν πολλέ θετικέ επιλογέ. πρέπει όμω σε περίπτωση κρίσεων να κάνουμε και τι δύο επιλογέ, των δύο λογιών επιλογέ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Κύριο Πόρτα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εμείς οι βουλευτές έχουμε τη δύναμη να αποφασίζουμε από μόνοι μας. Για τους μισθούς μας, παραδείγματο χάρη, ή για την πρόσληψη κάποιων ατόμων. Μεταξύ 11 και 12 αποφασίσαμε ότι θα παίρνουμε πάνω, 3.000 ε, ευρώ παραπάνω. Επίσης, Ψηφίσαμε για τις δαπάνες για γραφεία, για τα γραφεία μας, επιδοτήσεις, επιδόματα μάλλον, τα έξοδα μετακίνησης κτλ. Ε, λοιπά. Έχουμε λοιπόν ε, τη δυνατότητα να παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις. Σας ρωτώ λοιπόν το εξή. Τελικά χρησιμοποιήσαμε τις δυνάμεις της εξουσίας αυτές ή κάναμε κατάχρηση αυτών. Τις χειριστήκαμε με σοφία ή ήμασταν ανίκανοι να αντισταθούμε στους πειρασμούς που συνδέονται με τις εξουσίες που έχουμε. Φοβούμαι ότι δεν δείξαμε σοφροσύνη. Και τελικά η συζήτηση που κάνουμε σήμερα δεν έχει να κάνει με νούμερα, έχει να κάνει με ηθική, έχει να κάνει με πολιτική. Είναι μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει να πει πάρα πολλά σε αυτούς στους οποίους είμαστε υπόλογοι. Δεν είμαι δημαγωγός. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική είναι χάσιμο χρόνου. Ούτε λέω ότι θα πρέπει να δουλεύουμε οι ευρωβουλευτές υπό το φως των κεριών. Απλά είπα ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί. Αυστηροί και με τους δικούς μας, με, με τους εαυτούς μας όταν λαμβάνουμε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τα χρήματα και δι' αυτά τα οποία παίρνουμε εμείς. αλλάζουν τα πράγματα υπό τις παρούσες συνθήκες. Ε, δεν λέω ότι αυτοί που ε, δεν ταξιδεύαν business, παρόλο θα πρέπει να αρχίσουν να ταξιδεύουν business. Έχουμε το στένος να ψηφίσουμε έστω υπέρ του παγώματος κάποιων δαπανών. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν βουλευτές που δεν σταματούν να υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει περιορισμό ε, μείωση των μισθών, μέτρα λιτότητα, ε, περιορισμό συντάξεων μισθών, αλλά όχι όταν του αφορά αυτό βέβαια. Για την Ευρώπη των Ελευθεριών και τη Δημοκρατία, Άντρεασεν, για ένα λεπτό, κύριε κυρία Άντρεασεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αύξηση του 2,3% του προπολογισμού που ζητά το Κοινοβούλιο θέτει ένα αμφιβόλο το αίσθημα ευθύνη του Βλέποντας τις διάφορες δαπάνες βλέπει κανείς ότι υπάρχουν πολλές που αυξάνουν κατά 50 με 100% χωρίς κάποια λογική δικαιολογία. Αρχές της Ολομελίας ζήτησε από το Κοινοβούλιο να αναβάλει την ψηφοφορία για την έκθεση Φερνάντες λόγω ελήψεως ακριβών πληροφοριών και δαπανών για το Ευρωπαϊκό Σπίτι της Ιστορίας και για συγκρόμενα συμφέροντα. Αλλά το αίτημά μου καταψηφίστηκε. 2,5 εκατομμύρια ήδη πληρώθηκαν, εκταμιεύθηκαν χωρί να υπάρχουν αρκετέ ε, πληροφορίε. Φαίνεται οι ευρωβουλευτέ είναι πρόθυμοι να κινούνται στο σκοτάδι και να δίνουν χρήματα του φορολογουμένου χωρί να θέτουν τα σωστά ερωτήματα. Δεν μπορώ παρά να ρωτήσω τον Βρετανό Πρωθυπουργό να το πω να δεχθεί τίποτα από άλλο από σημαντικό, σημαντική μείωση όλου του κοινοτικού προβλησμού του 2012 και ελπίζω το Κοινοβούλιο να υποστεί τι μεγαλύτερε περικοπέ. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους μη εγγεγραμμένους. Συν... Συνάδελφος Χάρτονγκ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, τι να πω σε ένα λεπτό για τον προπολογισμό του 2012 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ε, μπορώ να πω πολλά, αλλά αρκετά. Δεν υπάρχει όραμα. Αποτελεί μόνο ε, κενές φράσεις, αποτελείται από κενές ε, φράσεις χωρίς προευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σπατάλες. Για παράδειγμα, στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ε, είναι τεράστια ο υπολογισμός του κόστους και η Επιτροπή συμμετέχει, η Επιτροπή Προπολογισμού συμμετείχε στην Επιτροπή ε, Εποπτείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι τελείως ε, απαράδεκτο. Ο κ. Λαμασούρ είπε ότι θέλει να διαθέσει την εντολή του προς αυτή την κατεύθυνση ε, και το κόμμα μας θα τον καλεί να το κάνει αυτό. Ελπίζω τον επόμενο χρόνο να περιοριστούν οι σπατάλες και να σταματήσουν. Εν μεταξύ θα εξακολουθώ να ελέγχω και να προειδοποιώ εξ του πολίτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση με τους άλλους εγγραμμένους αγορητές, ξεκινώντας από την κυρία Ματέρα για δύο λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον εισηγητή του προσωρινού προπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου, τον κύριο Φερνάντες, διότι κατάφερε να ισοσκελίσει τα αιτήματα της Γενικής Γραμματείας με τις προτάσεις του Επιτρόπου Λεβαντόφσκι σχετικά με τη συγκράτηση των διοικητικών δαπανών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το μήνυμα που αυτό το Κοινοβούλιο θέλει να δώσει είναι αυτό της υπευθυνότητας διατηρώντας τα αιτήματα για αυξήσει των κονδυλίων κάτω από το επίπεδο του πληθωρισμού μια στιγμή δυσκολίας για τα δημοσιονομικά των κρατών μελών. Εύχομαι το Συμβούλιο που θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση του εισηγητού για τη μείωση του μέγιστου του κεφαλαίου 5 για τους σκοπούς χρηματοδοτήσεως πολιτικών υπέρ των νέων να εκφραστεί ε, θετικά. Θεωρώ ότι το να διστάζουμε συμπληρωματικού φόρους για υποστήριξη της απασχόλησης των νέων τώρα ε, δεν τυχάνει υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να πατήσουμε τον γκάζι για να πετύχουμε τους βασικούς στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 και να επαναπροθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη η οποία θα βελτιώσει τη δυνατότητα των νέων μας να έχουν κατάρτιση και εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Το λόγο δίνουμε στον κύριο Φάρμ, τον κύριο Φάρμ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ οι συνάδελφοι που είναι αντίθετοι με την Ένωση είναι σαφές ότι θέλουν να περικόψουν και τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Αλλά όλα βασίζονται σε ένα λαϊκισμό. Αυτό είναι, που είναι το πιο σημαντικό είναι να δείξουμε ότι είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θεωρούμε ότι πρέπει να εξετάσουμε τις διοικητικές δαπάνες τώρα. Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε με αυτή την έκθεση να μην αποδεκτεί μία εξέλιξη που οδηγεί σε μία αύξηση του προϋπολογισμού. Σε περιστάσεις όπου εθνικοί προπολογισμοί, τα εθνικά δημοσιονομικά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και οι πολίτες ε, υποφέρουν από τη λιτότητα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε με κάθε σοβαρότητα. Τώρα όσον αφορά το θέμα αυτό, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που στο Κοινοβούλιο, ε, κάνουμε πραγματικές περικοπές. Και συμφωνώ με αυτό που είπαν πολλοί συνάδελφοι, θα πρέπει όμως να κινηθούμε με μεγαλύτερη στατηγική και γι' αυτό υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες ε, από την πλευρά των σοσιαλδημοκρατών για να γίνει πραγματική στατηγική αναθεώρηση των δαπανών του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι και εμείς στα σοβαρά κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει να εργαστούμε, να επανεξετάσουμε τα πάντα. Κάτι άλλο που ήθελα να πω. Αυτός ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας που αναφέρεται. Ε, πολλοί αμφισβήτησαν αυτό το θέμα, αλλά είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου ασχοληθεί με τέτοιο πρόγραμμα. Βεβαίως αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά το έργο αυτό, το πρόγραμμα αυτό ε, χρειάζεται να επανεξεταστεί. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφάνεια, ε, να φαίνεται ξεκάθαρα πού πάνε οι δαπάνες και να υπάρχει υπευθυνότητα, έλεγχος. Ε, οι πράσινοι, οι σοσιαλδημοκράτες και οι συγητής θα πρέπει να συμφωνήσουν ούτω ώστε να ψηφίσουν τις τροπολογίες μας για να καταλήξουμε σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το σχέδιο αυτό για τον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας να καταλήξουμε μια απόφαση πριν πλήρη διαφάνεια. Κύριε Φάρ, ε, υπάρχουν δύο αιτήματα με γαλάζια κάρτα να υποβάλουν ερωτήσεις εσάς. Δεχόσαστε. Καλώς. Χάρτονγκ, ε, το πρώτο ερώτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς τον συνάδελφο. Τι, έχει, τι είναι λάθος ε, με τον λαϊκισμό. Ε, οι βουλευτές είναι η φωνή του λαού, ακριβώς. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε Χάρτονγκ, ο λαϊκισμός σημαίνει συνήθως ότι δεν λαμβάνουμε αναλογικά και σοβαρό, σοβαρά τα πράγματα. Ότι δεν έχουμε μια στρατηγική. Γιατί το ουσιώδες που θα πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έναντι του φορολογούμενου και να ελέγξουμε ρεαλιστικά την πολιτική εξόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απλά τα πράγματα ασφαλώς για όσους δεν θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι να λαμβάνουμε τις ευθύνες μας, είναι λαϊκισμός. Ευχαριστώ ο κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. να ρωτήσω το εξή. Το Προεδρείο κατέθεσε μία πρόταση και προφανώς η έκθεση αυτή θα οδηγήσει σε κάποιες περικοπές, σε κάποια οικονομία για την εφαρμογή του προϋπολογισμού του 2010. Σε σύγκριση με αυτήν βλέπουμε 11% αύξησης και 174, 174 ε, εκατομμύρια ευρώ. 43 εκατομμύρια για έπιπλα, 30 εκατομμύρια για κοινοβουλευτικούς βοηθούς, 70 εκατομμύρια για ε, εκστρατείες ενημέρωσης. Χρειάζεται πραγματικά να συνεχίσω. Mr. Portas, you don't need... Όχι κύριε Πόρτας, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε και βασικά συμφωνώ μαζί σας και εγώ θα ήθελα να πάμε παραπέρα δεν με ικανοποιεί η αύξηση του 2,3%. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα. Ήταν όμως αυτό αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμού και του Προεδρείου και γι' αυτό καταθέσαμε πολλές τροπολογίες για να αναθεωρήσουμε την πολιτική δαπανών του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι μπορούμε να το πράξουμε αυτό με καλύτερη διαχείριση και πραγματική προσπάθεια για να γίνουν οικονομίε. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα διοικητικά έξοδα. Και εκεί θα ακούσουμε ασφαλώ ποιε είναι οι προτάσει του κυρίου Πόρτα. Σα ευχαριστώ. Χάγκλουντ για 1,5 λεπτό. Ο Χάγκλουντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ διεξάγεται μια συζήτηση ζωηρή, αλλά τα είχαμε κουβεντιάσει αυτά και πέρσι. Και όπως είπε και ο συνάδελφος από τους σοσιαλδημοκράτες, είναι καλό να υπάρχει μια στρατηγική εξέταση της μελλοντικής προσέγγισης. Με τέτοιο ζήτημα μπορεί κανείς να κάνει διαγωνισμό ποιος είναι ο πιο λαϊκιστής, δυστυχώς. Όμως πρέπει να επανεξετάσουμε τις δαπάνες μας. Και αυτό να το δούμε μακροπρόθεσμα. Εμείς, σαν φιλελεύθεροι και πέρσι και φέτος, προτείναμε οικονομίες. Και είμαστε μεταξύ εκείνων που ήθελαν περικοπές. Περισσότερα από αυτά που αρχικά προβλεπόταν. Ευχαριστούμε του τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Αυτό ο οίκος ευρωπαϊκής ιστορίας. Νομίζω είναι καλό να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται περί μακράς διαδικασίας που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη ε, θητεία του Κοινοβουλίου. Και ε, ίσως θα έπρεπε να διεξαχθεί μια ψηφοφορία, να δούμε ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, να ακουστεί η φωνή του καθενός. Νομίζω ότι δεν κερδίζουμε τίποτα να κάνουμε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού. Αντιθέτω, να σκεφτούμε σοβαρά πού μπορούμε να κάνουμε περικοπέ. Ευχαριστώ. Βαντάλεν για ένα λεπτό. κύριε Βαντάλεν. Πρόεδρε, στην παρούσα οικονομική συγκυρία θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κάνει καταρτήσει ένα προπολογισμό περιορισμένο και δικαίω ο εισηγητής ε, αναφέρει αυτά που αναφέρει. Δυστυχώ όμω δεν προχωράει αρκετά. Οι προτάσει ε, τώρα είναι να έχουμε προπολογισμό με αύξηση 2,3%. Αυτό δεν συνάδει με αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ούτε με αυτά που επιθυμεί το Συμβούλιο, που θέλει να περιοριστεί οι δαπάνες. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε οικονομίες. Μπορούμε να κάνουμε οικονομίες έχει αποφασιστεί ενδεχομένω στο παρελθόν να οικοδομηθεί αυτό ο οίκο ευρωπαϊκή ιστορία. Μπορούμε όμω να αλλάξουμε αυτή την απόφαση, να την αναστείλουμε. Αυτό το project το οποίο καταναλώνει δισεκατομμύρια. Και νομίζω ότι κάθε μήνα λαμβάνουμε πολλές χιλιάδες ευρώ για αποζημίωση. Χωρίς να ε, εξηγούμε λεπτομερώς αυτά τα έξοδα. Να κοιτάξουμε λοιπόν και να ελέγξουμε ε, αυτά τα έξοδα. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να γλιτώσουμε πολλά χρήματα προκειμένου να κάνουμε πιο πολλέ οικονομίε. Σα ευχαριστώ. Φερέιρα, για ένα λεπτό κύριο Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί μίλησαν για τους μισθούς των βουλευτών και τα επιδόματα που παίρνουν. Θα πρέπει να πω όμως ότι εμείς είχαμε καταψηφίσει ε, τα σχετικά με τους ε, βουλευτές του Κοινοβουλίου γιατί μεταξύ άλλων είχαμε διπλάσια αύξηση των ε, μισθών αλλά και για μια άλλη θεμελιώδη αρχή τη σύνδεση του μέσου μισθού των βουλευτών και του μέσου μισθού αυτών που εκπροσωπούμε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοιο χάσμα μεταξύ των εκπροσωπούντων και των εκπροσωπουμένων. Είναι θέμα ηθικής. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις, αλλά εμείς να είμαστε προστατευμένοι από τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Πράγματι, πολλοί θέλουν οικονομίες, αλλά για τα πολιτικά κόμματα είναι πολύ πιο ευνοϊκή η μεταχείριση. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η έκθεση για τον περιβολισμό του Κοινοβουλίου για το έτος 2012 υπογραμμίζει και σωστά την αναγκαιότητα συγκράτησης των δαπανών ο συμβιβασμό που επετεύθη φαίνεται να είναι αποδεκτό με την, μείωση τη αυξήσεω στο 2,3%. Άρα λιγότερο του πληθωρισμού. Άρα με μια θεωρητική οικονομία. Όμω ακόμα απόρα έχουμε από τα αιτήματα του Επιτρόπου για τον Περιπολογισμό. Και θα θέλαμε, ε, ήθελε να συγκρατήσουν τι ανάγκε του σε, σε αύξηση μόνο το 1%. Και κάποιοι όπω το Συμβούλιο κατάφεραν να το κάνουν αυτό. Α αφήσουμε εκτό τα θέματα που αφορούν αυτή την αύξηση. Πιθανότατα δικαιολογείται τι ε, μεγαλύτερα καθήκοντα και ευθύνε μετά τη Λισαβόνα. Να μιλήσω τώρα για αυτόν τον οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορίας. Στην Επιτροπή Προπολογισμών αναφέρθηκαν τρελά νούμερα όσον αφορά αυτό τον οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορία για την υλοποίηση και διαχείριση του οίκου αυτού. Είναι παράξενο, παράδοξο αυτή τη στιγμή να μπορούμε καν να σκεφτόμαστε να επενδύουμε δεκάδε επί δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για ένα πρόγραμμα, έργο που είναι αμφιβόλου χρησιμότητα εκτό τόπου και εκτό χρόνου. Ευχαριστώ. Βέρτμαν για 1,5 λεπτό. Κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, παρούσα ε, κρίση στα κράτη-μέλη για το έτος του 2012 ε, περιορίζει τον προϋπολογισμό του για το 2012 είναι κάτι που πρέπει να απενέσουμε. Γιατί αυξάνονται οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, η οικονομία αποτελεί την βασική μας αρχή το Κοινοβούλιο στον τομέα του, του προσωπικού ε, προβαίνει σε ε, οικονομίες και περιορίζει τα αντιπορικά έξοδα. Υποστηρίζω ιδιαίτερα την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να συνεχιστεί η πολιτική για το περιβάλλον του Κοινοβουλίου. Επίσης τονίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί την αρχή αυτή της οικονομίας. Ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε ευρέως. Άρα καλωσορίζουμε το γεγονός ότι ο ότι γίνονται, αποτρίβονται τα σχετικά κονδύλια στο project. Και εκεί αναμένουμε μείωση των εξόδων και θέλουμε πλήρη διαφάνεια σε όλα τα σημεία. Σας ευχαριστώ. για Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι για μα ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό κάθε χρόνο αποτελεί μία πρόκληση. Αφενός θέλουμε να κάνουμε οικονομία, αφετέρου θέλουμε αποδοτικά να δαπανίσουμε τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μα. και νομίζω ότι στον τομέα της αποδοτικότητα μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνουν προτάσει βελτίωση σε ό,τι αφορά ε, τους βουλευτές, τους βοηθούς τους, προκειμένου να βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητα του Ευρωκοινοβουλίου αφετέρου από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά ε, έχουμε απέναντί μας ε, υπουργούς που έχουν ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό στο γραφείο τους, στα εθνικά κράτη-μέλη και τα σχετικά, τη σχετική χρηματοδότηση, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εξηγήσουν ε, στο εσωτερικό της χώρας τους, στην πολιτική την ευρωπαϊκή. Και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε υπεύθυνοι για να προσεγγίσουμε τον λαό προκειμένου να εξηγήσουμε τι αποφασίζουμε κάθε ημέρα. Οι νέες αρμοδιότητες στην ενέργεια, στην εξωτερική πολιτική, στην, στην πολιτική ανταγωνισμού, στην πολιτική για το περιβάλλον, για τα κοινωνικά ζητήματα είναι θέματα που προαπαιτούν την ύπαρξη των σωστών μέσων. Θα πρέπει να κοιτάξουμε που υπάρχουν δυνατότητες οικονομίας. Δεν τίθεται θέμα. Όπου μπορούν να γίνουν οι οικονομίες θα πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι για κάποια βασικά θέματα είμαστε ε, όλοι υπεύθυνοι να καθορίσουμε πόση δουλειά έχουμε και όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στην διακριτική ευχαίρεια των βουλευτών. Γιατί είναι καθοριστικής σημασίας να συνεχίσουμε να έχουμε καλή επικοινωνία. Ε, κύριε Ρούμπικ, ο κύριος Γκέιερ για 1,5 λεπτό παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούγοντα τη συζήτηση που διεξάγεται για τον οίκο τη Ευρωπαϊκή Ιστορία, μου φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο δύο είδη βουλευτών. Αυτοί που είναι υπέρ του προπολογισμού, που συμμετέχουν σήμερα εδώ στη συζήτηση και είναι κριτικοί έναντι τη ε, διαδικασία αυτή, και όλοι οι υπόλοιποι που είναι υπέρ. Το πρόβλημα είναι ότι ε, ανάγεται αυτό το θέμα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει να κάνει τίποτα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι το κόστος ε, για τον οίκο αυτό είναι 107 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ από την Daily Telegraph ε, δεν μπορώ παρά να καλέσω κάποιον να κοιτάξει τα έγγραφα αυτά και η διαφάνεια που απαιτείται από τους βουλευτές ε, να υπάρξει και στο σημείο αυτό, γιατί θα ήθελα να ελέγξω αυτά τα έγγραφα που μιλούν για τέτοιους αριθμούς, αστρονομικά ποσά. Είναι σκοπός ε, να... Χρειάζεται μάλλον το Κοινοβούλιο ένα μουσείο. Όχι, σίγουρα όχι. Γι' αυτό και για τους σοσιαλδημοκράτες υπάρχουν οι εξής δύο γραμμές. Ότι θέλουμε ένα business plan για το project αυτό και κατά δεύτερον ότι θέλουμε μελέτη αντικτύπου και όλα αυτά θα πρέπει να έχουν διευκρινιστεί. Και κάτι τρίτο που θα ήθελα να προσθέσω, ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις σε ό,τι αφορά το Info Center και τον Νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ε, για ένα λεπτό. Øh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να δω κάτι πάνω σε αυτό το μουσείο τον οίκο αυτό. Διότι είναι καλό το Κοινοβούλιο να μπορεί να χειριστεί, να διαχειρίζεται αυτό το μουσείο. Καλό θα ήταν όμως να υπάρχουν καλύτερες δομές για τις επισκέψεις στο Κοινοβούλιο και στις Βρυξέλλες και, στο, και το Μουσείο Ευρωπαϊκής Ιστορίας να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα του συνόλου. Σημαντικό ποσοστό της ομάδας είναι υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας όμως συμφωνούμε και με αυτά που είπαν οι σοσιαλιστές. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο ανοιχτή προσέγγιση για να ξέρουμε πού ε, διατίθεται τα χρήματα, ποια θα είναι η οικονομική κατάσταση, το κόστος της διαχείρισης, το μέλλον του μουσείου. Είναι καλή ιδέα όμως η ιδέα αυτή καθευτή και την υποστηρίζω. Πρέπει να ξέρουμε όμως τι συνεπάγεται οικονομικά. Και αυτό μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Είσαστε ακριβή το χρόνο παρόλο το ότι είχατε ένα λεπτό. Για δύο λεπτά ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ. Ε, Ιδίωσε αυτή τη στιγμή είναι επίμαχο θέμα ο προπολογισμό, ιδίω αυτή τη χρονική συγκυρία. ενηρία και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι όλοι είχαν την δυνατότητά τους να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ακούσαμε όλες αυτές ε, τις απόψεις ε, και αυτή είναι και μία από τις σημαντικότερες, ε, τα, τα μεγαλύτερα ισχυρά σημεία του Κοινοβουλίου ότι ακούγονται οι απόψεις όλων. Σίγουρα είναι δύσκολη η κατάσταση από οικονομικής πλευράς και οποιαδήποτε αύξηση δεν θα, ληφθεί, δεν θα δοθεί με θετικό μάτι. Και συμφωνώ σε έναν βαθμό, αλλά τελικά σε τελική ανάλυση έχουμε μια αύξηση 2,3% ενώ ο προπολογισμό αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,8%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να δει και το πλαίσιο και την κατάσταση σε κάθε μια από τις 27 χώρες μέλη. Η δική μου χώρα, παραδείγματος χάρη, πλήττεται αυτή την περίοδο. Με τον Επίτροπο Ρέν είχαμε μια συνάντηση μόλις πριν, ο οποίος ευτυχώς ήταν πάρα πολύ καλός μαζί μας και σίγουρα υπό την παρούσα συγκυρία ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα ε, όταν μιλάμε για αύξηση. Ίσως αν είναι κάτω βέβαια από το επίπεδο του πληθωρισμού κάτι μπορεί να καταλάβει. Έχουμε να κάνουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, πράγματι με τη συνθήκη της Λισαβόνας αυξάνονται οι αρμοδιότητές μας ε, και το θέμα είναι το εξής. Πριν ολοκληρώσω να προσθέσω. Όλα αυτά μας φέρνουν κατά νου αυτό το οποίο πολύ συχνά λέει ο πρόεδρος Μπαρόζο πρέπει να γίνει μια πλήρης και ειλικρινή συζήτηση για τους ίδιους πόρους και ίσως και για τα ομόλογα για έργα, τα project bonds. Διότι όσο μεγαλύτερη και ανεξάρτητη είναι η χρηματοδότηση που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο λιγότερα θα ζητάμε από, την Ευρωπαϊκή, ε, από τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή και τη σύσταση του Μπαρόζου. παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ εδώ το κόμμα που είναι πιο πολύ υπέρ της Ευρώπης από τη χώρα μου, την Ολλανδία. Και επειδή πιστεύω στην Ευρώπη τόσο πολύ, είμαι επικριτικό σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή τη δύσκολη ε, χρονική συγκυρία θα πρέπει να κάνουμε μεγάλες οικονομίες και δεν συμφωνώ με την αύξηση του προπολογισμού και μου προκαλεί κυρίως έκπληξη ο αρχικός προϋπολογισμός ε, τον οποίο κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας άνω του 5% αύξηση μου προκαλεί έκπληξη που δεν είναι εδώ θα ήθελα να είναι εδώ να το υπενθυμίσω το σημείο 6 του ψηφίσματος όπου ζητάμε από τις υπηρεσίες να χτενίσουν τον προπολογισμό για να κοιτάξουν πού μπορούν να γίνουν οικονομίες. Και θα ήθελα να του ζητήσω πριν από 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους να το έχουν και ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη για να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε οικονομίες. Και τέλος θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους που είναι υπέρμαχοι της Ευρώπης να μην δίνουμε όπλα στα χέρια των πολέμιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ο λαός ε, που επικαλούνται ε, θα υποφεληθεί από μια ισχυρή Ευρώπη. Εδώ για δύο λεπτά παρακαλώ. Θέλω να συγχαρώ τον ε, εισηγητή Φερνάντες και να ευχαριστήσω τον προλαλήσαντε γιατί ήταν πολύ εύστοχα αυτά που είπε. Πράγματι είναι πιο λιτός ο προπολογισμό με βάση και αυτά που ζήτησαν Συμβούλιο και Επιτροπή. Διατηρείται το όριο του 20%, άρα ε, συμφωνούμε με αυτή τη συμφωνία κυρίων, μάλλον τηρούμε τη συμφωνία κυρίων παρότι δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες ε, κομματικές ε, τοποθετήσεις νομίζω, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Παραδείγματος χάρη θέλουμε όλοι να υπάρχει καλύτερη νομοθετική παραγωγή, θέλουμε να τηρήσουμε τις νέες προτεραιότητες στη συνθήκη της Λισαβόνας όπως μας ζητείτε, θέλουμε να είμαστε πιο επαγγελματικοί ε, και όπως ε, μας ζητούν. Μας ζητούν να έχουμε περισσότερες αίθουσε συνεδριάσεων, καλύτερη επικοινωνία, καλύτερα δίκτυα πληροφορική. Πώ θα τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. Δεν χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να πληρωούμε και τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει για θέματα ακινήτων. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πάψουμε να τα χρηματοδοτούμε αυτά, αλλά αυτό δεν λειτουργεί έτσι και αν είμαστε υπεύθυνοι πρέπει να το δεχθούμε, έτσι. Έτσι δεν είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νεολαία, εδώ πράγματι είναι ένα επίμαχο θέμα. Ε, αλλά ποτέ δεν πρέπει να είναι επίμαχο γιατί είναι αναγκαιότητα. Έχουμε στη χώρα μου, παραδείγματο χάρη, 50% νεανική ανεργία. 100 εκατομμύρια ευρώ στην πολιτική για την νεολαία δεν, για την νεολαία δεν θα λύσουν τα προβλήματα. Τουλάχιστον όμω θα ανταποκριθούν στι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την κατηγορία 5 μέχρι την κατηγορία 1α η μεταφορά των 100 εκατομμύριων ξέρω ότι θα ε, δημιουργήσει ε, κάποιες αντιρρήσεις και έχουμε και την διαδικασία του περιπολισμού. Είμαστε όμως ένας ζωντανό οργανισμός και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της στιγμής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο, ε, πιο κατεπήγον θέμα από το να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων και είμαι βέβαιος ότι όλοι έχετε την ίδια προτεραιότητα. Α, και κάτι άλλο. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ του σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάνερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον συντάκτη τη εκθέσεω, τον κύριο Φερνάντε, για την έξοχη δουλειά που έκανε. Αυτή η άξιση του 2,3% είναι πιο εύκολο να γίνει αποδεκτή, είναι πιο εύκολο να δικαιολογηθεί από ότι το 5,2% που προτάθηκε από το Προεδρείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ασκήσει αυτοκριτική όσον αφορά τον προπολογισμό του. Αυτό συμπεριλαμβάνει αυτή η έκθεση, αλλά πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε οικονομίε και στι ε, μικρολεπτομέρειε. Παραδείγματο χάρη, ε, η οικονομία για τα απορριπαντικά. Ε, ίσως θα πρέπει να έχουμε και ψηλότερους στόχους από ότι να οικονομούμε μόνο στο σαπούνι και στα απορριπαντικά. Κατά διάρκεια του έτους το Κοινοβούλιο ψήφισε ούτω ώστε η διπλή σύνοδος του φθινοπόρου να γίνει μία σύνοδος, μία μόνο εβδομάδα. Αυτή η μηνία μετακίνηση θα μπορούσε να σταματήσει και αν το κάνουμε αυτό θα κάνουμε σημαντικές οικονομίες. Ευχαριστώ. Πολύ κυρία Μάνερ. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο τέσσερις συνάδελφοι από ένα λεπτό ο καθένας γιατί έχουμε καθυστέρηση το χρόνο μας. Ε, θα πάρει το λόγο τώρα ο κύριος Ζέμκε. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε το λόγο. Αν δούμε τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δούμε ότι οι, δαπών, οι δαπάνες για τις μεταφορές είναι σημαντικές και θα εξακολουθήσουν να είναι. Είμαστε 27 ε, χώρες, μετακινούμαστε από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο, από τις χώρες μας στις Βρυξέλλες κτλ. Και ξέρουμε ότι το κόστος ε, μετακίνησης των βουλευτών και των άλλων Ευρωπαίων εργαζομένων σίγουρα και υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να εξοικονομήσουμε ε, λίγο παραπάνω. Σίγουρα ταξιδεύουμε, ταξιδεύουμε πολύ αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο για τα αεροπορικά εισιτήρια πρέπει να πληρώνουμε το ίδιο με αυτούς που χρησιμοποιούν σπαραδικά μόνο το αεροπλάνο. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κάποια συμφωνία με τις αεροπορικές εταιρείες αφού χρησιμοποιούμε τόσο πολύ ε, τις αεροπορικές μεταφορές. Ξέρω ότι πολλά υπουργεία έχουν ε, σημαντική έκπτωση στη 20% και... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η έκθεση την οποία συζητούμε αφορά το θέμα 17 και 18 για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, όπου και προτείνεται να δημιουργηθεί αποθεματικό για τα περαιτέρω έξοδα του project αυτού, του σχεδίου αυτού. Στο άρθρο 10α αναφέρονται τα αποθεματικά για τα καταπήγοντα έξοδα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το project. Άκουσα ότι είπαν οι συνάδελφοι, οι προλαλήσαντες οι οποίοι και ε, ανέφεραν ότι τα κόστος για τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας ε, έχει υποτιμηθεί κατά πολύ. Καταλαβαίνω δεν καταλαβαίνω μάλλον τα άτομα ε, εκείνα τα οποία εμένουν σε αυτό το σχέδιο σε, περιο... σε εποχές κρίσης. Ξέρω ότι η... δημόσια εικόνα της Ευρώπης θα πληχθεί καθότι θα θεωρηθεί αυτό σπατάλι. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω το project αυτό να το ξανασκεφτούμε. Το Βαμπένοβα έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα από την έκθεση να υπογραμμίσω το εξής. Τη φιλοδοξία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τις οικονομίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εποχές όπου πολλοί κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χάσει τους μισθούς τους, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός συνοδεύεται από αυστερούς δημοσιονομικούς κανόνες προκειμένου να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε, για παράδειγμα, σε θέματα ηλεκτρονικής διοίκησης ή χρήσης ε, βιντεοδιασκέψεων. Να τα υποστηρίξουμε όλα αυτά προκειμένου να κάνουμε οικονομία και να μην χρησιμοποιούμε και ε, με φυσικούς πόρους και στο χαρτί για παράδειγμα να κάνουμε οικονομία. Είναι βασικό. Να μην επηρεάσει αυτό την εργασία μας, για παράδειγμα στις επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ ε, τον Σάρφο Φερνάντες ε, για την εξαιρετική εργασία του καθώς επίσης και την εξαίρετη συνεργασία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Γραμματείας της Επιτροπής ε, για την εξαίρετη συνεργασία. Όπως είπαμε και στη συζήτηση, ε, μια, ε, υπήρχε η πρόταση του 5,2% για το 2011 και φτάσαμε σε ένα συνολικό ε, καθεστώς το οποίο ε, έχει αύξηση 2,3%. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντική ε, η πρόβλεψη μεταφοράς 100 εκατομμυρίων για προγράμματα υπέρ της νεότητος, πολιτική την οποία θεωρεί κατά προτεραιότητα πολιτική για το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί με την εργασία για όλους τους νέους Ευρωπαίους και την κινητικότητα και την εκπαίδευση αφορούν σημαντικά στοιχεία για τον επόμενο επόμενο χρόνο. Ελπίζουμε ότι και μέσα από την δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων θα βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των πόρων. παρακαλώ, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πολύ καλή έκθεση. Επίσης, ε, όλοι οι βουλευτές που πήραν το λόγο τόνισαν τα προβλήματα και τις λύσεις. Η μόνη όμως καλή λύση είναι να μην αναζητεί ο καθένας ε, ελλείμματα, προβλήματα, με νυφαλαιότητα και αντικειμενικότητα να δούμε τα θέματα. Το Ενεκτικό Συνέδριο έχει ζητήσει και έχει ήδη ε, διεξαγάγει εξωτερικό οικονομικό έλεγχο και δείχνει αυτό ότι γίνονται καλές και σωστές οικονομίες. Γι' αυτό ελπίζω να υποστηρίξετε την τροπολογία μου, να ελέγχετε και έξωθεν το κοινοβούλιο. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα. Και είπε και Γιώχαν Κάμπ εδώ ότι αυτό το κόστος στο ε, μέλλον θα πρέπει να αναφερθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη του ότι διανύουμε μια δύσκολη οικονομική συγκύρια και είναι αρκετά περίπλοκες και οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου μας στο δυνατόν πιο αποδοτικό τρόπο, έτσι ώστε οι δαπάνες για το 2012 να αυξηθούν κατά 2,3%, δηλαδή χαμηλότερα από τον, από τον πληθωρισμό. Αυτό νομίζω θα ήταν ένα πολύ θετικό μήνυμα. Το όλο που χρειαζόμαστε είναι πιο, αυστηρές, πιο αυστηρούς κανόνες παρακολούθησης των δαπανών. Ένα σύστημα, αν θέλετε, πολυετούς παρακολούθησης και νομίζω πως εδώ καθένας από εμά θα πρέπει να κάνει προσπάθειες για να εξορθολογήσουμε την διοίκηση του Κοινοβουλίου και για να χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπινους πόρους με αποτελεσματικό τρόπο. Ελπίζω λοιπόν πως έτσι θα εξοικονομήσουμε χρήματα για το φορολογούμενο και θα μειώσουμε τις δαπάνες του Κοινοβουλίου. Ε, και τώρα θα κλείσει τη συζήτηση ο εισηγητής μας ο κύριος Φερνάντες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να τονίσω πόσο σημαντικό είναι πως τα διοικητικά έξοδα, οι διοικητικές δαπάνες όλων των ευρωπαϊκών οργάνων φτάνουν στο 6%. Δεν υπάρχει κανένας προϋπολογισμός σε κανένα κράτος μέλος που να είναι τόσο μικρό ποσοστό τα, οι διοικητικέ δαπάνε του συνολικού προπολογισμού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εδώ έχουμε την πρωτιά. Και έχουμε νέες αρμοδιότητες, έχουμε 27 κράτη-μέλη. Έχουμε την συνθήκη της Λισαβόνας που έχει τεθεί σε ισχύ. Και έχουμε βέβαια και τους επιπλέον 18 ευρωβουλευτές. Τι σημαίνουν όλα αυτά, πώς αυξάνουμε και τις δαπάνες μας και Ταυτόχρονα βέβαια αληθεύει πως έχουμε μια πραγματική μείωση ε, στον προϋπολογισμό αυτό γιατί είμαστε κάτω από το ρυθμό αύξηση του πληθωρισμού. Δεν γίνεται λοιπόν αυτόματα μια αναπροσαρμογή. Βέβαια χρειαζόμαστε να εγκριθεί στο Συμβούλιο με ομοφωνία, αλλά αυτό που στέλνουμε εμείς είναι ένα μήνυμα. Στα διοικητικές δαπάνες λοιπόν στο 5 που αναφερόμαστε στα 380 εκατομμύρια ευρώ, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να εισάγουμε αυτές τις πρωτοβουλίες για τον αυστηρότερο έλεγχο. Τώρα, για τους μισθούς των ευρωβουλευτών, εμείς δεν μπορούμε να τους αναπροσαρμόσουμε κατά βούληση. Είναι το Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την ε, χάραξη της μισθολογικής μας, αν θέλετε, πολιτικής. Είχαμε μία πρόταση της τάξης του 0,9% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βρίσκεται και στον εσωτερικό κανονισμό και νομίζω ότι έχει να κάνει ε, με τις αποφάσεις του ΔΕΚΣ στο συγκεκριμένο τομέα. Επαναλαμβάνω όμως πως για όλα αυτά είναι απαραίτητη η έγκριση του Συμβουλίου. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να διαβάσουν το 323. Μια ερώτηση στον εισηγητή. Κύριε Φερνάντες, θα δεχτείτε μια ερώτηση από τον κύριο Πόρτας. να έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ο, ο, ο Κύριε Φερνάντες, για το θέμα αυτό των μισθών των ευρωβουλευτών, νομίζω και είναι προφανές αυτό κατά τη γνώμη μου, πως το Κοινοβούλιο μπορεί να αναλάβει τέτοιου είδους πρωτοβουλίο και μπορεί να προτείνει μια αναθεώρηση ε, του καταστατικού στο σημείο αυτό για τους ίδιους τους βουλευτές και νομίζω ότι αυτό έχει εγκριθεί και εδώ και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με το να κάνουμε εμείς αυτή την αναθεώρηση. Πιο συγκεκριμένα θα σας πω πως είναι ο μισθός ο οποίος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι υπόλοιπε δαπάνες σχετικές με τους μισθούς εξαρτώνται άμεσα από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε εμείς εδώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως επιβεβαιώνει ο κύριος Πόρτας, δεν είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου ο καθορισμός των μισών των βουλευτών. Οπότε δεν έχει νόημα ένας τέτοιος ε, προϋπολογισμός να μιλάει για πάγωμα των μισών. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε μια πρόταση τροποποίησης του καθεστώτος των βουλευτών. Επίσης θα είχε νόημα να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Το άρθρο 64 και ο κανονισμός 31. Αυτό που δεν έχει νόημα είναι να ε, προσπαθούμε εδώ στο Κοινοβούλιο να λέμε ότι οι βουλευτές αυξάνουν τους μισθούς τους όταν αυτό ε, δια νόμου απαγορεύεται. Αλλιώ είναι δημαγωγία και λαϊκισμός. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έληξε η συζήτηση εδώ και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης. Είναι η έκθεση του κυρίου Ιβάν προστασία των οικονομικών συμφερόντων